Επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση. Για τη μέση διάταξη ζητεί κάποιο το λόγο. Ποιο, ο κύριο Έπινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σα επίσης την προσοχή σε μια περίπτωση διαφθορά στην τσεχική δημοκρατία. Ο κύριο Ντέιβιτ Ράτ, ένα κυβερνήτη βοημό ε, ε, από τη βοημία, μάλλον συνελήφθη, ήταν υπουργό υγεία διότι έφυγε από τον τόπο που διέπραξε το έγκλημα και τον πιάσανε με 7 εκατομμύρια τσεχικές κορώνες. Άλλοι 7 επίσης συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για επεξαίρεση και είναι κοινοτικά χρήματα. Ε, χρήματα από τα ταμεία, σύμφωνα με εκθέσεις στις εφημερίδες, από καλές πηγές, αξιόπιστες. Επίσης είχε κρύψει ο κυβερνήτης αυτός περίπου 30 εκατομμύρια κορώνες, 1,2 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από το πάτωμα στη βίλα του. Αυτό το σκάνδαλο συνεχίζεται στη τσεχική δημοκρατία και εφόσον αφορά δημόσια χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία, ε, θα ήθελα να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει τι συμβαίνει, να το μάθουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Διότι πρέπει να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη, να δώσουμε απαντήσεις. Και θα ήταν χρήσιμο να μας απαντήσουν τι τρέχει. Θα πρέπει να τεθεί το θέμα αυτό στο σημείο, σαν σημείο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης ε, συνεδρίασης. Ευχαριστώ συνάδελφε. Μας επιστήσετε και την προσοχή. Δημοσιεύματα του τύπου έχει ζητήσει το λόγο. Αλλά σας, ε, και άλλοι συνάδελφοι, παρακαλώ σύντομα όμως γιατί είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat eh, v současné době. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα, ο κύριος Ράτ, που είναι βουλευτής ε, στη Τσεχική Βουλή και πρώην κυβερνήτης ε, της Βοημίας, ε, κρατείται ε, για παθητική δωροδοκία. Είναι σημαντικό αυτό, είναι σοβαρό αυτή τη στιγμή ε, είναι στη φυλακή ένας ε, βουλευτής, βεβαίως και ο τύπος αντιδρά. Την άλλη εβδομάδα θα ε, αρχίσει η δικαστική διαδικασία και πιστεύω ότι η περίπτωση αυτή θα ερευνηθεί και θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Μάλιστα. Ο κύριος Πίπερ. Uh, Πρόεδρε. Έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και προτείνω να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Όλα αυτά τα σημαντικά να τα πούμε άλλη φορά αργότερα. Τώρα όμως να ψηφίσουμε. Ναι, και εγώ αυτό θα πρότεινα. να περάσουμε στην ψηφοφορία. Αλλά ε, για την τσεχική περίπτωση ο κύριος Γκάιερ. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να παρατείνω τη διαδικασία ούτε να αναφερθώ στην τσεχική υπόθεση και να λάβω θέση, αλλά να κάνω μια γενική παρατήρηση. Άτυπα, έχουμε ήδη συζητήσει λίγο για τις τροπολογίες του κυρίου Πίπερ στη γνωμοδότηση του κυρίου Βον. Αν ε, προσφέρονται όλες αυτές τις τροπολογίες να ψηφιστούν εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σημειώνω ότι η κυρία Χιούμπνερ, πρόεδρος της Περιφερειακής Πολιτικής, έχει την ίδια άποψη ότι δεν μπορούν έτσι να ψηφιστούν όλες οι τροπολογίες του συναδέλφου Πίπερ γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ούτε την ποιότητα ε, των τροπολογιών που ε, θα άρμοζε σε δική μας γνωμοδότηση και θέλω να κάνω παρατηρήσει γενικέ. Βεβαίω, κάθε βουλευτή έχει δικαίωμα να κάνει παντού τροπολογίε. Το βλέπουμε και στην έκθεση Μαρινέσκου που έχει βγει από την ημερήσια διάταξη σήμερα. Έχουν έρθει συνάδελφοι με διάφορε τροπολογίε. Συνάδελφοι που δεν έχουμε δει ποτέ εδώ στην Επιτροπή. Εντάξει, δικαίωμά του, μεγιά του, με χαρά του. Το θέμα όμω είναι εάν κάθε τροπολογία που κατατίθεται επί τη ουσία ταιριάζει σε κάθε έκθεση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ότι είναι εκτός θέματος, εκτός τόπου και χρόνου. Υπάρχουν άλλα που είναι εντός και άλλα που είναι φαιά ζώνη. Κοινώ γκρίζα. Αυτή θέλω να ξεκαθαριστεί και για να μην σας ε, ταλαιπωρήσω, ούτε ζητώ να ληφθεί κάποια απόφαση τώρα, αλλά θέλω να πω εξ ονόματος της ομάδας μου ότι υποστηρίζουμε πλήρως την κυρία Χίμπνερ που μας έστειλε την άποψή της σήμερα το πρωί και να το ξαναδούν οι συντονιστές παρακαλώ αυτό. Να βρούμε κάποια διαδικασία και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να ασχολείται με τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια καθήλυν και επί της ουσίας. Ήθελα να τα πω αυτά και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να το σκεφτούν και να προβληματιστούν ενδεχομένω και στην ψηφοφορία να τηρήσουν ανάλογη στάση. Ευχαριστώ. Δύο είναι τα πράγματα και δεν θέλω να τα αναμίξω. Θέλω να πω στον κύριο Έπινγκ ε, ότι συμφωνώ να το ελέγξουμε αυτό το θέμα ε, της Τσεχίας και να το κλείσουμε εδώ και ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία, στη μερίσια διάταξή μας δηλαδή. Και ως πρόεδρος σας έχω στείλει την επιστολή της κυρίας Χιούμπνερ που είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και εκφράζει την ανησυχία η κυρία Χιούμπνερ ότι ορισμένες τροπολογίες που θα ψηφίσουμε ενδεχομένως να μην είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Και δεν θα μπορούσαν να είναι. Θέλω να σας πω το εξή σχετικά με αυτό. Εχθές και στην Επιτροπή μας αλλά και σε προηγούμενη συνεδρίαση των συντονιστών και γενικότερα συζητήσαμε τι γίνεται με άλλες επιτροπές που μπαίνουν στα δικά μας χωράφια, α πούμε ειδική έκθεση για τις απαιτήσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα, γιατί μου είπατε και εσεί εχθέ ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής να ε, υπερασπιστώ τα συμφέροντά μας και ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και παντού όπου ε, θίγονται ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και η Περιφερειακή Επιτροπή ε, επιτρέπεται αλλά και θα έπρεπε να γνωμοδοτεί. Και εγώ θα αγωνιστώ γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μία τάση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να περιοριστούμε στην εκτονιστέρων έλεγχο των οικονομικών. Όχι, δεν είναι αυτή μόνο η δουλειά μας και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και τους εαυτούς μας και την Επιτροπή. Ε, διαπιστώνω και στη διάσκεψη των Προέδρων ότι έρχεται γι' αυτό ε, στο παρελθόν δεν το οξύναμε ως σύγκρουση και σε ό,τι αφορά το άρθρο 50 και 51 του κανονισμού, αλλά τώρα κανονικά θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες, να δούμε τις τροπολογίες επιμέρους για να ελέγξουμε αν έχουν οικονομικές επιπτώσεις ή όχι. Αλλά και οι μετεβατικές λεγόμενες περιφέρειες έχουν οικονομικές επιπτώσεις και το θέμα της δυσκολίας ε, της εφαρμογής ε, των πολιτικών και της απορρόφησης κονδυλίων έχει σχέση με αυτά που συζητούμε παράδειγμα η τροπολογία 35 Φερρυπίν. Δεν καταλάβαμε ε, ότι οι τροπολογίες που λέτε κύριε Γκάιερ δεν είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Πρόκειται πολύ περισσότερο για ε, πολιτική υπόθεση και αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ψηφιστούν. Αυτά για τη διαδικασία. Τώρα θέλετε να κάνουμε συζήτηση για τον κανονισμό, για το ποιε απολογίες ψηφίζονται και ποιε όχι. Εγώ θα πρότεινα να ψηφιστούν όταν δεν είναι προφανές αν είναι δική μας αρμοδιότητα ή όχι. Αυτό είναι πολιτική αξιολόγηση. Τι να κάνουμε. Να τις ψηφίσουμε λοιπόν και θα διαμορφωθεί η πολιτική ε, άποψη και μετά θα δούμε τι θα γίνει και με την ε, ε, Περιφερειακή Επιτροπή. Γιατί δεν αφισβητεί κανεί την Επιτροπή Ρέγγι ότι είναι καθήλυνα αρμόδια και επί τη ουσία και εμεί γνωμοδοτούμε. Αυτά είναι, αυτή είναι δική μου προσωπική άποψη. Θέλει κανεί το λόγο, κύριο Πίπερ. Όχι, δεν θέλω συζήτηση να γίνει τώρα. Να πω μόνο στον κύριο Γκάιερ ότι μπορώ να καταλάβω την παρατήρησή του υπάρχουν τροπολογίες που και εγώ δεν ήμουν σίγουρος, ε, αλλά το ήλεγξαν οι υπηρεσίε της Γραμματείας. Και για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αγαπητέ συνάδελφοι, ε, την περασμένη εβδομάδα προτείναμε στον κύριο Βον να τα ελέγξει ε, κάποια ζητήματα που είναι αβέβαια και κρίσιμα και είμαστε και διατεθειμένοι να αποσύρουμε τις τροπολογίες και ήρθε κατηγορηματική η απάντηση ότι καμία από τις δικές μου τροπολογίε δεν είναι παραδεκτή στην Επιτροπή Ελέκτου Προπολογισμού. Ε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, ότι όλε μου οι τροπολογίε είναι απαράδεκτε και δεν ψηφίζονται. Μάλιστα, δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Μήπω να ψηφίσουμε, σα παρακαλώ. Το σημείο 12 λοιπόν. Η έκθεση Βόν. ein. Άρθρο 2, η τροπολογία 32, ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, σας παρακαλώ, για την 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι, πέρας. εψηφίστε ψηφίστε τότε. Okay. Ja, ja. Äh, es ist, äh, äh, ich war etwas zu schnell. Α, βιάστηκα. Δεν ξέρω, ψηφίσανε όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, 15-11 εγκρίνεται χωρίς αποχές. Η 33 ψηφί υπέρ, παρακαλώ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 36 όχι 35 διορθώνει ο πρόεδρος 35 κατά αποχές εγκρίνεται η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία υπαρθμών 37 υπέρ Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη τροπολογία υπαρχών 37. Ψηφίσατε όλοι. Όλοι και όλες. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 38 ψήφιπε. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές, επειδή είναι σαφές παρακαλώ να το επαληθεύσουμε, είναι η τροπολογία 19, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 19. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, ήταν σαφές μάλλον, εγώ δεν το είχα δει, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 20 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 39 Πε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 Πε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τη 43 η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ένας υπεράριθμος. Έδειξε το ηλεκτρονικό σύστημα ότι ψηφίζει ένας σοσιαλιστής και δημοκράτης παραπάνω από τους δικαιούς. Μάλιστα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Εντάξει. Τροπολογία 44 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 44 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Hat Ψηφίσατε όλοι. Τώρα είναι ένας λιγότερος. Τι θα γίνει. Πέρασε. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Η 45 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και πάλι κατά πλειοψηφία. 48 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 48 αρχίζει τώρα, σας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πάλι περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Συγγνώμη. Ψηφίζει ένας παραπάνω. Α, και τώρα ένας λιγότερος. Μπορείτε να τα βρείτε σας παρακαλώ. Εγώ δεν ψηφίζω λέει ο κύριος Γκάιερ. Εγώ έχω βγάλει την κάρτα μου. Ναι, αλλά και κάποιο άλλο συνάδελφο, ο κύριο Κάλφιν, τώρα είναι ένα λιγότερο δηλαδή. Θέλετε να ψηφίσετε, κύριε Κάλφιν. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 16-10 με δύο αποχές. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει ελεγχό. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 21. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 50 ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51 παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό δεν ήταν σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 52. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 54 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 54. Check is geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 55 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 56, η 57 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56 και 57 μαζί αρχής ψηφοφορία Hat jeder abgestimmt? Der Check ist geschlossen. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίψετε. 22 καταπίπτει. Η τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. 58. Τι λέει εδώ, καταπίπτει αν εγκριθεί 1 η οποία έχει αποσυρθεί όμως. Άρα ψηφίζουμε την 58. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Υπέρ κατά οι ε, 4 ε, αποχές εγκρίνεται. Η 59 υπέρ ε, κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 59. Παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Α, ναι, Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία είναι 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται επίσης 63 επέρ, κατά άποχες εγκρίνεται 64 υπέρ κατά άποχες ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 64 αρχίζει τώρα ψηφίσατε όλοι πέρασε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 Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 76. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 77 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 και 24 και 25. Μαζί, όχι. Χωριστά. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 έχει αποσυρθεί όπως και η 6 ερχόμαστε στην 80 ψήφι υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 80. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς, ζητώ συγγνώμη. Μητροπολογία τροπολογία 7, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81, υπέρ. Κατά αποχές και αυτό θέλει έλεγχο. 81 παρακαλώ, αρχίζει ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 8 έχει αποσυρθεί όπως και η 9. Ερχόμαστε στην 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 έχει αποσυρθεί πάμε στην 84 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την 84 ηλεκτρονικά. Νικά. Πέρασε. Εγκρίνεται 18 υπέρ κατά. 85 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ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 Haben alle Kolleginnen Kollegen. Ναι, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 17 υπέρ, 11 κατά. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά. Μήπως θέλει και το λόγο ο συνάδελφος. Όχι. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία. Ακολουθεί η έκθεση του συναδέλφου Γιάννης Γκάιερ. Ψηφίζουμε. Άρθρο 5, παράγραφος 6. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. 6. Ψήφι υπέρ. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι για την έξι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαρθμόν 1. Ψήφι πέρα. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Τροπολογία 7 καταπίπτει και 20 και ερχόμαστε στην τροπολογία 8. Ψήφι π Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθυμών 9. Ψήφι π Της 9. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθυμών 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές δεν είναι πάρα πολύ σαφές σας παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 12 ψηφίζουμε αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέρας. όντως ήταν μικρή διαφορά 13 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται ήταν η τροπολογία παρθών 12 αυτή έτσι ωραία 21 καταπίπτει, όπως και 22 και πάμε στη 13. Ψηφίπε Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν φαίνεται ακριβώς τι γίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 14. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 ψήφιπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 καταπίπτει 16 16π, Κατά. Άποχες. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 16 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται η ένα ψήφι περ κατά απόχες εγκρίνεται η συσυμβαστική παριθμό 2 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η τροπολογία 17 κατά πίπτη 2, 18 ψηφίζουμε την 3 ψηφί υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπάρχουν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 4 παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να ε, ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά Γιάννη Προχωρούμε επόμενη έκθεση. Das 10, äh, Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Η συγητής είναι ο κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη. Και ψηφίζουμε. Το άρθρο 7, παράγραφο 3, τροπολογία 15, ψήφι Κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 15 Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 καταπίπτει. 17 ψηφιπέ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά εποχές Εγκρίνεται. Η 9. Ε, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ του πρώτου τμήματος στις 10. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 1 καταπίπτει. Η 2 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε τη 2 παρακαλώ γιατί δεν κατάλαβα τι έγινε. Ηλεκτρονικά πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία εδώ και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία και τελειώνει. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατάργηση του κανονισμού. Τάδε. Συγητής Καταλήν Σόριν Ψηφίζουμε Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4 έχει αποσυρθεί. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθμών 7. Για στιγμή. τι λέει εδώ, ψηφίζουμε μόνο εφόσον η 5 απορριφθεί. Η 5 εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτουν η 7 και οι 8. Έτσι δεν είναι. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, ψηφίζουμε την 7 και την 8 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 αποσύρθηκε η 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 11 Ηλεκτρονική Abstimmung geschlossen. Εγκρίνεται. 12 και 13 μαζί επε κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε μαζί τις δύο 12 και 13. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνει. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 και 16 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 και 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο της γνωμοδότησης ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Πέρασε. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα. Προπολογισμό του 2013 εντολή για τον τριμερή διάλογο. Συντάξει νομοδότηση είναι ο Κρίστοφερ Φιέλνερ. Μία τροπολογία έχει μόνο. μόνο ένα ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το σύνολο της νομοδότησης τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Α, όχι ακόμα. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα τελειώνει. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Φιέλνη. Και ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της Ιλιάνα Ιβάνοβα καινοτόμα και μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία παριθμών τρία υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτό υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 8 αρχίζει τώρα ψηφίσατε όλοι ε, ναι πέρασε απορρίπτεται σαφώς η υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης αρχίζει τώρα. Ηλεκτρονική Abstimmung Σαφές το αποτέλεσμα και συγχαρητήρια στην κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαν οι ψηφοφορίες για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ μεγάλη πειθαρχία. 10 στα 10, μπράβο σας, με τόνο. Και από χρόνο πάμε πολύ καλά και ερχόμαστε αμέσω στο επόμενο θέμα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ισπανία. Συγγνώμη, έχουμε τίποτα άλλο πριν. Α, κάτι ξέχασα. Oh, no, no, sorry. Yeah, yeah. Μάλιστα. Ξέχασα τίποτα γιατί σε μένα η μερίστη διάταξη λέει αντιπροσωπεία κοντ στην Ισπανία. Η δική έκθεση για την αλία μου λένε. Έτσι λέει. Αλλά ας δούμε πρώτα το θέμα της Ισπανίας και μετά την αλία είναι ενδιαφέροντες οι καιροί και το πλαίσιο γενικά και το πολιτικό στην Ισπανία. Αφενό υπάρχει νέα κυβέρνηση που κάνει πολύ μεγάλε προσπάθειε για να προετοιμάσει και να φτάσει στους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την εξυγίαση του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα ε, κοιτάμε και στο παρελθόν τι έγινε με τα κοινοτικά κονδύλια, γιατί από την Επιτροπή μας επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι θέλουμε να τα κοιτάξουμε ε, εκτενέστερα. Ε, το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον σε συνεργασία με τους Ισπανούς συναδέλφους, την Ισπανική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία μας και θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα αυτό το σημείο. Head of delegation is the colleague Derek. Ο Derek Vaughan ε, θα είναι ο πρόεδρος αντιπροσωπείας. Θέλει κανείς το λόγο για αυτό το θέμα της αντιπροσωπείας στην Ισπανία. Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, die Kollegin Ayala Sender, bitte schön. Συνάδελφος Ayala, παρακαλώ. Ινές, θέλεις να μιλήσεις για αυτό το θέμα της αντιπροσωπείας στην Ισπανία. Όχι. Α, ο κύριο Στάς λέει όχι. Δεν θέλει. Είναι Νέσα Μάλιστα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω κάτι εγώ. Είδα ότι από τους ντόπιου συναδέλφους, ο συνάδελφος Σαλβαδόρ Γαρίγα εδώ εμφανίζεται, δεν ξέρουμε ποια ιδιότητα, διότι θα ενδιαφέρονται ακόμα τρεις συνάδελφοι να συμμετέχουν που είναι μέλη της Κοκομπού πρώην και νυν κοντ. Κάποιοι ντόπιοι βουλευτές θέλουν να συμμετάσχουν και είναι μέλη της Επιτροπής μας σε ορισμένες συνεδριάσεις. Λοιπόν, ο κύριος Γκαρίγα ως τι εμφανίζεται. Εντάξει, είναι Ισπανός συνάδελφος, αλλά υπάρχουν και τρεις άλλοι που είναι μέλη της Επιτροπής μας. Από τη Βαλένσια, από τη περιφέρεια μου. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω. Βλέπω ότι στο πρόγραμμα τουλάχιστον προβλέπονται συνεδριάσεις με τους προέδρους των αυτονόμων περιφερειών και τους αντίστοιχους αρμοδίους ε, για τη διαχείριση των κονδυλίων, που είναι οι εμπειρογνώμονες και οι ειδικοί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν επιβεβαιωθεί όλες αυτές οι επισκέψεις και οι συναντήσεις και να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι είναι γεγονός ότι άλλαξε η κεντρική κυβέρνηση, ε, η ομοσπονδιακή όπως τα λέγατε στη Γερμανία, αλλά σε ορισμένες περιφέρειες υπάρχουν νέες κυβερνήσεις ενώ αλλού όχι. Στην ε, Βαλένθια και στην αυτόνομη περιφέρεια εκεί δεν έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Ε, θα μας ε, ενδιαφέρει να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί στο πρόβλημα που βρίσκουμε πάντα μπροστά μας ε, την πάγια αυτή η κατάσταση για τη δήλωση του αρμοδίου και αντιστοίχου υπουργού φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί αυτό ένα από τα προβλήματα που πάγια θέτουμε είναι τα προβλήματα μεταξύ της κυβέρνησης και των περιφερειακών κυβερνήσεων και τέλος να πω ότι στο πρόγραμμα εμφανίζεται συνάντηση με τους εκπροσώπους ε, του οργανισμού του κοινοτικού στο Αλικάντε. Πώς έτσι. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν επεσήμενε τίποτα. <laughs> Γιατί θα πάμε εσύ στο Αλικάντε ολόκληρο απόγευμα εκεί με τους υπευθύνους του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ja, Also die erste Frage η πρώτη ερώτηση νομίζω έχει εύκολη απάντηση. Τα μέλη της αντιπροσωπείας ε, αναφέρονται εδώ και έχετε στη διάθεσή σας τα έγγραφα. Ο Ντέρεκ Βον ε, είναι κεφαλής και τον ορίσαμε εμείς Εγώ στις 19 μόνο θα είμαι στη Μαδρίτη, δεν μπορώ να πάω στην περιφέρεια, θα πρέπει να γυρίσω στις Βρυξέλλες. Και τα μέλη από την εκάστοτε χώρα ε, μπορούν να συμμετέχουν στην ε, ερευνητική των πραγμάτων αποστολή. Οι Ισπανοί συνάδελφοι μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Να με διορθώσει η γραμματεία εάν δεν έχω σωστή ενημέρωση είναι εκτό της ποσοστώσεως οι ντόπιοι συνάδελφοι. Το άλλο θέμα με το οργανισμό στο Αλικάντε δεν μπορώ να το απαντήσω, το είχαμε συμφωνήσει. Θα προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω. Μπορείτε να απαντήσετε εσείς ίσω από τη γραμματεία. Να καλέτε. Mm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. So it was, uh, Μάλιστα. Δύο συνάδελφοι το ζήτησαν. Ο κύριος Τάμας Ντόιτς και ο κύριος Ρούμπιχ θέλησαν να επισκεφθούν τον οργανισμό στο Αλικάντε. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή, μια που θα είμαστε εκεί, να κοιτάξουμε και τον οργανισμό αυτό. Και αν δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια από πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου, είναι και ένα παράδειγμα καλή διακυβέρνηση. Δεν πάμε μόνο εκεί που υπάρχουν προβλήματα, πάμε και βλέπουμε και του οργανισμού που λειτουργούν καλά. Είμαστε που είμαστε στην περιοχή, γιατί να μην πάμε. Ο κύριος Γκάιερ και μετά η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στη σύνθεση της αντιπροσωπείας και στην παρουσία του συναδέλφου Γκαρίγκα εδώ; Πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι ακριβώς, πήγαμε στην ε, Ιταλία εκεί που είχαν γίνει σεισμοί και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον και ντόπιοι βουλευτές ε, από την περιφέρεια εκεί που δεν ήταν μέλη της Επιτροπής μας, ούτε πλήρη, ούτε αναπληρωματικά, ούτε τίποτα. Και τότε τους είπαμε, αφού το είχαν συζητήσει οι συντονιστές ε, επί ότι δεν μπορούμε να τους δεχτούμε στην αντιπροσωπεία μας. Γιατί ενδεχομένως τα αποτελέσματα και τα πορίσματα μπορεί να ήταν τελικά δυσάρεστα ή να μην ικανοποιούσαν πλήρως περιφερειακές αρχές και μπορεί να έφεραν αντιμέτωπους τους βουλευτές εκεί με ζητήματα και ερωτήματα. Εγώ συμφωνούσα τότε και αποθάρρυνα τους βουλευτές που δεν ήταν μέλη της Επιτροπής μας να συμμετάσχουν για την αποστολή και στην Ούμπρη, όπως σας είπα. Και κανονικά δεν τους δεχόμασταν στο παρελθόν. Και τώρα θα πρέπει να βρούμε και πάλι μια διαδικασία που να ισχύει πάγια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον συνάδελφο Γκαρίγα Πολιέδο, τον ξέρω από την Επιτροπή Προπολογισμών. και συντονιστής του ΕΛΚ μάλιστα και ικανός και άξιος. Αλλά αν πούμε ότι εδώ κάνουμε εξαίρεση, έτσι θα ενθάρρυνα και συναδέλφους από τη δική μου πολιτική ομάδα συμμετέχουν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, είτε θα βρούμε μια ρύθμιση για όλους και θα λέμε περιορίζεται η συμμετοχή ε, στα πλήρη και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μας, είτε το ανοίγουμε και ε, όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλά έχω και εγώ πιστούς. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάγια, για την πρακτική του παρελθόντος δεν ξέρω εγώ τι γινόταν. Εγώ προσανατολίστηκα στους ε, κανόνες που ισχύουν τυπικά και εξ όσων γνωρίζω δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κανένα. Μπορούν να το συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες ε, και προσωπικά, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα αυτά που μας λέτε. Κυρία Γκρέσλε, ο συνάδελφος Γκαρίγα μέχρι πρόσφατα ήταν ένα πνευματικό μέλος και θα το λύσουμε πολύ γρήγορα με την Ισπανική Αντιπροσωπεία, αν παραμένει απληρωματικό μέλος ή όχι. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα, γιατί μέχρι τις προάλλες ήταν ένα πραγματικό μέλος. Και μέχρι τώρα ισχύει αυτή η πρακτική όντως, μόνο μέλη πλήρη αναπληρωματικά. Αν έχει αλλάξει η Επιτροπή, καλώς. Αν έρθει ξανά στην Επιτροπή μας αναπληρωτής να τον πάρουμε μαζί μας, αλλιώς όχι. Να ρωτήσω κάτι για τον οργανισμό, γιατί δεν πρόσεχα τι λέγατε. Ποιος οργανισμός είναι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς στο Αλικάντε και προσκαλούνται εκεί σε μια συνομιλία. Να πω δυο λόγια. Δεν έχουμε δώσει εμείς απαλλαγή γιατί δεν παίρνει χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αλλά καλό θα ήταν να επισκεπτόμαστε όλους τους οργανισμούς και να μπουν και όλοι οι οργανισμοί στην απαλλαγή. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίβαχο με το Συμβούλιο. Αν θέλετε να δείτε τι εστί ευημερία και ευμάρια, πρέπει να πάτε εκεί. 40 εκατομμύρια ευρώ έχει έσοδα από ε, το, την πίσνα αυτή με τα σήματα Δηλαδή αρμέγουν κανονικά τη βιομηχανία και αυτά τα λεφτά δεν τα βλέπει κανείς. Γιατί το διαχειρίζεται εσωτερικά ο οργανισμός. Και έχει έτσι και πολύ αξιοπρεπή γραφεία στις Βρυξέλλες, για να μην πω πολύ τελή. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε την ε, ευημερία και την ευμάρεια στην πράξη, να πάτε. Εγώ δεν ξέρω από γεωγραφία εκεί είναι κοντά, αλλά αν υπάρχει ευκαιρία να πάμε. γιατί είναι πραγματικά αγκάθι αυτός ο οργανισμός και μας πονάει και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν αλλά να είμαστε και σωστά προετοιμασμένοι. Καλώς. Λοιπόν, αν μπορούμε να επισκεφτούμε, μπορούμε. Είναι 160 χιλιόμετρα. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί, τους προσκαλούμε όμως γιατί είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Και πάλι τώρα ζήτησε φυσικά το λόγο είναι σαν Γιάλα. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις. Για τον κύριο Γκαρίγα. Δεν είναι αναπληρωτής. Έχει φύγει από την Επιτροπή μας. Και όπως πολύ ωραία εξήγησε ο κύριος Γκάιερ, αν θεωρείται ο κανόνας είναι ότι δεν ταξιδεύουν, είναι ντόπιοι, είναι εκεί οι άνθρωποι. Είναι από τη Βαλένσια. Εντάξει, ο κύριος Γκαρίγα έρχεται πολύ για τον οργανισμό του Αλικάντε είναι αυτόνομος όπως ξέρει η κυρία Γκρέσλε, αυτό χρηματοδοτείται από τα εμπορικά σήματα και τα διπλώματα τεχνίας. Εγώ ούτε ξέρω τι γίνεται, ούτε έχω πάει, αλλά έχουμε ένα απόγευμα και θα έρθουν να μας συναντήσουν εκεί Και αντί να συναντάμε αυτούς, εγώ θα προτιμούσα να δούμε επιτόπου στη Βαλένθια διάφορα έργα και προγράμματα που έχουν εντοπιστεί προβλήματα. Αν θέλουν να έρθουν να συναντηθούμε, να κάνουμε μια συζήτηση, μια εξέταση, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το να πάμε, να έρθουν από την Αλικάντε στη Βαλένθια να μας συναντήσουν, αυτό είναι fact-finding mission, είναι διερευνητική ε, αποστολή. Εκτός του ότι αυτό χρηματοδοτείται αυτός ο οργανισμός, είναι εκτός θέματος. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα η κυρία Γκρέσλε να τον ελέγξουμε, αλλά από θέμα επιμελητίας και χρόνου ρωτούσα. Και οι συνάδελφοι που είναι στη Βαλένσια, δικοί μας συνάδελφοι ντόπια μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάποιες συζητήσεις για να μας βοηθήσουν να δούμε κάποια προγράμματα, κάποια έργα πιο ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε. Ε, έχουμε και στη Σεβίλη οργανισμό. Και άλλο στην Ισπανία, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Αλλά τον θυμάμαι πολύ καλά γιατί έχουν 40 ή 45 υπαλλήλους και 70 ή 79 ε, συμβούλου στο Εποπτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό είναι παράδειγμα οργανισμού. Δεν θυμάμαι ποιος οργανισμός είναι. Δεν ξέρω πόσο σφιχτό και πιεσμένο είναι το πρόγραμμα. Αλλά από τότε που είμαι τουλάχιστον εγώ μέλος εδώ στην Επιτροπή, είναι η πρώτη φορά που πάμε στην Ισπανία. Αν είχαμε χρόνο να καλέσουμε και τη δεύτερη αυτή υπηρεσία, το δεύτερο οργανισμό για να ασχοληθούμε και μαζί τους. Αλλά για το θέμα του Αλικάντε οπωσδήποτε και επιγόντω αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με. Δύο παρατηρήσει, λέει ο πρόεδρο. Εξ όσων γνωρίζω από άλλε επιτροπές, πώς έχει η κατάσταση. Συνάδελφοι που δεν είναι μέλη των εκάστοτε επιτροπών, αλλά είναι βουλευτές της χώρας, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν. Αλλιώς θα έπρεπε να εθετήσουμε την πρόταση του κυρίου Γκάιερ να το ε, ανακοινώσουμε. Εγώ δεν θέλω να το διατυμπανίσω. Η κυρία Γκρέσλι τοποθετήθηκε σωστά για τον κύριο. Κλείσουμε εδώ το σημείο. Να το κανονίσουν οι πολιτικές ομάδες. Το δεύτερο είναι το θέμα του προγράμματος. Ο χρόνος είναι σχετικά περιορισμένος όπως το βλέπω εγώ. Γιατί το βράδυ θα πρέπει να παίρνουμε το τρένο για τη Μαδρίτη. και δεν νομίζω να χωράει και άλλος οργανισμός στο πρόγραμμα. Να το κοιτάξει η γραμματεία όμως παρακαλώ. Ποιος άλλος έχει ζητήσει τώρα το λόγο? Äh, Κοιτάξτε, εγώ κατάλαβα, λέει ο κύριος Γκάιε, ότι ο οργανισμός του Ελικάντε θα έρθει να μας βρει στη Μαδρίτη. Και έχει και νόημα. Γιατί δεν μπορούμε, δεν προκάνουμε να πάμε στο Αλικάντο εμείς. Η κυρία Γκρέσλε μας είπε ότι έχουν γραφείο και στις Βρυξέλλες και αν θέλουμε να τους συναντήσουμε και να τους συζητήσουμε, τους καλούμε εδώ στην Επιτροπή και τελειώνει η υπόθεση αφού έχουν και γραφεία στις Βρυξέλλες. Έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα μετά από συνεννοήσεις και συζητήσεις που είχαμε κάνει στην Επιτροπή μας και έχουμε και κατάλογο προτεραιοτήτων από κοινού. Γιατί πάμε στην Ισπανία. Λοιπόν, παρακαλώ τους συναδέλφους να ξανακοιτάξουν το πρόγραμμα, να μην το ξαναανοίξουν. Του στείλα, ξέρετε τι σούπερ ιδέα κατέβασα. Να μην περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο την οργάνωση. Γιατί είναι και πολιτική η ατζέντα. Αλλιώ θα πρέπει όλα να τα δει από την αρχή η γραμματεία. Ευχαριστώ. Κύριε ε, ε, Γκάιερ, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα και ευχαριστούμε και τη γραμματεία που το προετοίμασε έτσι και το κατήρθησε. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Ορτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε δείτε. Διάφορα θέματα έχω εγώ να πω. Πρώτον, να πούμε ότι πάμε στην Ισπανία γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι θέλουν να επικεντρωθούμε στη Βαλένσια, αλλά υπάρχει και Ανδαλουσία και η Καστίγια Λαμάντσα. Δεν πάμε μόνο στην περιφέρεια της Βαλένσια. Επίσης, το παρελθόν, κανείς δεν είπε για την ΟΑΜΗ. Ο ΟΑΜΗ θα πάει στη Βαλένσια, όχι στη Μαδρίτη. Του Αλικάντε δηλαδή οι εκπρόσωποι θα έρθουν στη Βαλένσια, όχι στη Μαδρίτη. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Είναι πολύ χρήσιμο να επισκεπτόμαστε κάποιους ε, οργανισμούς επιτόπου, αλλά... Καλό είναι να δούμε τι είναι η Βαλένσια και η Περιφέρεια και η Ισπανία για να μην δαιμονοποιούμε κανέναν. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Αγιάλα, δυστυχώς δεν την ακούμε. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι πολύ θετικό να δείχνουμε κάποια πράγματα που λειτουργούν και κάποια άλλα που ενδεχομένω να δυσλειτουργούν. Έτσι δεν είναι. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι η επίσκεψη είναι στην Ισπανία, όχι μόνο στην περιφέρεια της Βαλένθια. Και στην Ανδαλουσία είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και στην Καστίγια Δαμάντσα. Δεν είναι αποστολή στην Βαλένθια. Ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη αυτή έχετε απόλυτο δίκιο. Η χώρα μέλος λέγεται Ισπανία. Ναι. Εκεί πάμε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ωραία. Σπουδαία, θαυμάσια. Δεν θα ήθελα να παραλείψω εδώ να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίασή μας και τον τμήματάρχη κύριο ε, Μαϊράτε. Ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας. Σας δίνω το λόγο για να μας ενημερώσετε από πλευράς δικής σας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω, θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη ενημέρωση, ένα briefing, ε, παρατηρήσεις για το πρόγραμμα, ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ και πάλι και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σπουδαία υποστήριξη. Well, thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, σας δώσαμε ένα briefing που είναι συνοπτικό. Κατά την επίσκεψη θα έχετε πολλές ευκαιρίες να συζητήσετε την εφαρμογή των ταμείων στην Ισπανία στο σύνολό τους. Αλλά να σας κάνω και μερικές γενικές έτσι, περιγραφές για το τι προβλέπει το πρόγραμμα. Σας θυμίζω ότι η Ισπανία παίρνει τα μεγαλύτερα ποσά από τα ταμεία αυτά. 170 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί στην Ισπανία από το 89. 4 με 5 δισεκατομμύρια πληρωμές γίνονται κάθε χρόνο. Άλλο σημαντικό τα ποσά αυτά τα διαχειρίζεται κεντρικά το Υπουργείο Οικονομικών αλλά υπάρχουν και 145 ενδιάμεσα σώματα τοπική αυτοδιοίκηση ή τίποτε άλλοι οργανισμοί. Στο παρελθόν, την προηγούμενη δηλαδή περίοδο, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις που ταυτίσαμε ιδιαίτερα ως προς τις δημόσιες προμήθειες, διότι ο σχετικός νόμος δεν συμφωνούσε με την κοινοτική νομοθεσία. Αλλά μειώθηκε ο κίνδυνος λάθους στις δοσοληψίες. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα και γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο και η Κομισιόν τα αναφέρουν. Αλλά γενικά η κατάσταση βελτιώθηκε τα περισσότερα προβλήματα σήμερα αντιμετωπίζονται. Η Κομισιόν έχει πάρει μέτρα ας πούμε διακόπτει τις πληρωμές πολλές φορές πέρυσι με 13 από αυτά τα ενδιάμεσα από τους ενδιάμεσους οργανισμούς απευθυνθήκαμε σε 13 και για το 11 9 σε 9. Βέβαια δεν μιλάμε μόνο για συστημικές ελλείψεις αλλά και για μεμονωμένα λάθη που δεν αφορούν το σύστημα στο σύνολό του. Υπά, γίνονται δημοσιονομικοί έλεγχοι τακτικά από την Κομισιόν και επίσης τακτικές συναντήσεις συντονισμού ώστε να είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπιστούν τα λάθη. Και επομένως μπορέσαμε να κάνουμε τμηματικές μερικές πληρωμές και με αυξημένη εγγύηση. Αυτό το δείχνουν και οι τελευταίοι δημοσιονομικοί έλεγχοι. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει τρεις επισκέψεις σε τρεις περιφέρειες. Γιατί αυτές, διότι ήταν εκείνες όπου το ελεγκτικό συνέδριο είχε ταυτίσει προβλήματα το 10. Και αυτό προτείνουμε αυτές τις τρεις περιφέρειες. Εν τω μεταξύ έχουν ληφθεί ορισμένα διορθωτικά μέτρα και η κατάσταση έχει βελτιωθεί, όχι τελείως τακτοποιηθεί, αλλά βελτιωθεί. Τέλος, στο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα συνάντησης με τις κεντρικές αρχές, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα την αρμόδια αρχή για τη διαχείριση αυτών των ποσών και ταμείων. Και έτσι μπορείτε να τους πείτε ό,τι θέλετε για τη διαχείριση. Την τρίτη μέρα θα συναντήσετε τις ελεγκτικές αρχές, είναι μία κεντρική αρχή, και θα μπορέσετε και εκεί να θέσετε ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ταυτιστεί από την Κομισιόν ή από το Ελεκτικό Συνέδριο. Να αυτά έτσι γενικά για το πρόγραμμα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε γιατί επέλτρεις περιφέρειες. Τώρα θέλουν μερικοί να χαλιάσουν οι νέες πρώτοι και καλύτεροι. Ευχαριστώ Ευχαριστώ και εγώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βοήθειά του στην προετοιμασία του προγράμματος και για τις εξηγήσεις του. Και θέλω να τον ρωτήσω στο συγκεκριμένο ζήτημα των ε, κρατικών προμηθειών και των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί, σε ποιο επίπεδο έχει ληφθεί η απόφαση. Γιατί υπάρχουν ε, επίπεδα τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βλέπει ότι χωρούν βελτιώσεις ε, στις δημοσίες συμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο επιδέχεται βελτίωση, αλλά πού διαπιστώθηκαν τα προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις, σε ποιο επίπεδο διακυβέρνηση. Ε? Ευχαριστώ. Άλλος. Κυρία Γκρέσλε. Τον γνωρίζουμε καλά τον κύριο ε, Μαϊράτε, γιατί ήταν μαζί μας και στην αντιπροσωπεία στη Λάκουιλα, εκεί που είχαμε πάει στους σεισμούς της Ιταλίας. Αν ε, συγκρίνουμε την Ιταλία με την Ισπανία, έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους, γιατί εδώ και 10 χρόνια είναι στα διαστατικά ταμεία επικεφαλής των ατασταλιών. Περισσότερο στην Ισπανία από ό,τι στην Ιταλία είναι... Ε, οι τις λειτουργίες και είναι πρόβλημα. Χαίρομαι που ακούω σήμερα ότι βελτιώθηκαν τα πράγματα, αλλά από πότε θα ρωτούσα και μάλιστα τι βελτιώθηκε. Γιατί εξακολουθούμε να βλέπουμε υψηλά ποσοστά ασφαλμάτων εδώ και 10 χρόνια και καιρό είναι και ο κύριος Μαριάτε να λάβει θέση. ποιε είναι οι βελτιώσεις, ποιε είναι οι ουσιαστικές βελτιώσεις και γιατί εδώ και 10 χρόνια με πραγματικά η όβια υπομονή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθεται και τα δέχεται όλα αυτά. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Άλλες, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Well, um, if I may on the... Κοιτάξτε, για το πρώτο θέμα για τις προμήθειες θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου από το τμήμα εποπτείας ελέγχου. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω τι διαπιστώσαμε για τις βελτιώσεις στην Ισπανία. Το 5 ταυτίσαμε τα πρώτα προβλήματα. Το 6 εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο ζητούσαμε από τις Ισπανικές Αρχές να βελτιώσουν τους ελέγχους και να διορθώσουν τα πράγματα στα συμβόλαια δημοσίων προμηθειών αλλάζοντας τα συμβόλαια και τη χρήση, τα κριτήρια επιλογής. Οι Ισπανοί εφάρμοσαν το σχέδιο το 7 και 8. Το ΔΕΝΕΑ 9 ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος διορθώθηκαν 2,5 δισεκατομμύρια εξοικονομήθηκαν από την ανάλυση όλων των συμβαλέων. Και μετά οι Ισπανοί έκαναν αλλαγές στην ομοθεσία τους για να... για να βελτιωθούν και άλλο τα πράγματα και το σημαντικότερο μέτρο που έλαβαν στο, στην προγραμματική περίοδο 7 με 13 είναι η συμπερίληψη μιας ρήτρα επιλεξιμότητας που απέκλειε τις μετατροπές των συμβολέων και για την τωρινή προγραμματική περίοδο δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει καμία παραβίαση. Αυτές που βρίσκουμε αφορούν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν από τη λήψη αυτών των μέτρων. Τι συμβόλαια αφορά αυτό το πρόβλημα όλων των ειδών συμβόλαια, όλων των Τα όρια που προβλέπονται δεν αφορούν τα προβλήματα αυτά. Όλα τα συμβόλαια αφορούν. Όλα. Σας κατευχαριστώ. Τι θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Ναι, για να απαντήσω αυτά που είπε η κυρία Κρέσλε. Είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς την Ιταλία με την Ισπανία γιατί τα δύο συστήματα διαφέρουν. Στο ελεγκτικό συνέδριο και τους ελέγχους του η Ισπανία και η Ιταλία εμφανίζονται συχνά γιατί είναι από τις χώρες που ωφελούνται περισσότερο από τεράστιες πληρωμές και γι' αυτό διαπιστώνουμε περισσότερα λάθη. Για την Ισπανία Υπάρχουν βελτιώσεις, δηλαδή υπάρχει ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα, οργανισμός που ταυτίζει τα περισσότερα λάθη. Αυτό δεν υπάρχει παντού. Και γι' αυτό αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και το κεντρικός αυτός οργανισμός που λέγεται η ΓΑΕ διασφαλίζει ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα όποτε πρέπει πριν γνωμοδοτήσει και εγκρίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν διαπιστω... ε, βελτιώσεις στην Ισπανία. Όλα τα αποτελέσματα από αυτό το Εθνικό Ελεγκτικό Σώμα τα στέλνει στην Κομισιόν και τα λαμβάνουμε υπόψη μας εμείς. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Και λίγη εδώ και αυτό το θέμα. Προσβλέπουμε δε στην επίσκεψή μας εκεί στην Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ. Πάει και αυτό το σημείο. Και ερχόμαστε στο επόμενο που είναι η ειδική έκθεση ε, για την απαλλαγή του 2011 για τον αλληλευτικό στόλο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Μάρτα Ανδρέασεν, για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίτλος μου είναι πώς συνέβαλαν τα ευρωπαϊκά μέτρα στην προσαρμογή του αλληλευτικού στόλου στις δυνατότητες που έχουμε. Και η απλή απάντηση είναι ότι τα μέτρα δεν έχουν συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Το ελεγκτικό συνέδριο έκανε μία αποτίμηση. Η κοινή αλληλευτική πολιτική προωθεί τη βιώσιμη λέει αλληλεία αλλά η μείωση της υπεραλίευσης δεν σημειώθηκε, δεν επιτεύχθηκε. Οι αλλιεύσεις μειώθηκαν κατά ένα εκατομμύριο τόνους, χάθηκαν 100.000 θέσεις εργασίας και τελικά 1,7 δισεκατομμύρια σπαταλήθηκαν από το 2002 στον παροπλισμό για τον παροπλισμό πλοιαρίων. Για την απαλλαγή λοιπόν του 11 πρέπει να δούμε ποια ευθύνη έχει η Κομισιόν για όλα αυτά. Καταρχάς δεν κατάφερε να, να μετρήσει ποια ακριβώς είναι η υπεραλίευση. Δεύτερον, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση, εφαρμογή των ελευτικών δικαιωμάτων. Τρίτον, δεν υπάρχει σαφής ορισμός των κριτηρίων επιλογής για τα πλοιάρια στα οποία εφαρμόζονται τα προγράμματα της Κομισιόν. Και τέλος, δεν πέτυχε να ελέγξει, να πετύχει, δεν πέτυχε την ενημέρωση των ε, καταλόγων των πλοιαρίων, των μητρώων. Γενικά συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά τις ξεπερνώ. Αρνούμε την απαλλαγή για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Δεν νομίζω ότι έχει πετύχει η μεταρρύθμιση και συστήνω η κοινή αλληλευτική πολιτική να πάψει να εφαρμόζεται εφόσον δεν προσφέρει τίποτα και πρέπει να αφαιθεί στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τρέσσα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου από το ελεγκτικό συνέδριο και αν υπάρχουν ερωτήσεις και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Ιβάνοβα, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος συναδέλφου Φέλνερ που χρειάστηκε να λείψει. Ευχαριστεί την κυρία Αντρέσεν για την έκθεσή της, καθώς και το συνέδριο για τις πληροφορίες που μας χορήγησε. Σας τον τους κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα. Ραϊόφ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια και το ελεκτικό συνέδριο. Είναι πολύ κρίσιμο το θέμα αυτό και επικριτικό και δικαίως. Γιατί πρόκειται για την κοινή αλευτική πολιτική της Ένωσης. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το ελεκτικό συνέδριο μας επισημαίνει πού πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε αυτό το μέσο να γίνει πιο χρήσιμο και ωφέλιμο για την κοινότητα. Και μια που είμαστε και στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, είναι και επίκαιρο το θέμα. Γι' αυτό και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, έχει σημασία έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και πάρα πολύ επίκαιρη γιατί ε, μπορούμε τώρα να ε, οξύνουμε κάποια ε, εργαλεία και μέσα. Συμφωνώ και ο δισηγητής με πολλές από τις εκτιμήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια εκεί που λέει ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πανεθνικοποίηση. Στην Αρμόδια Επιτροπή συζητούμε πάρα πολύ σκληρά και επώδυνες συζητήσεις για τις ποσοστώσεις ε, και τι θα σημάνει αυτό για τον αλλιευτικό κλάδο κάθε χώρα. Στη δική μου χώρα είναι όντως οδυνηρό γιατί εκείνοι που ασχολούνται με το περιβάλλον έχουν διαφορετική θεώρηση από εκείνους που προέρχονται από αλευτικές κοινότητες. Και υπάρχει μια διαμάχη και δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με επανεθνικοποίηση. Και όποιος μπορεί να αυξάνει το στόλο του θα τον αυξήσει και μετά θα αδειάζουν οι θάλασσες με τρόπο άτακτο και άναρχο. Αυτό μπορεί στην αρχή να ενισχύσει την αλληλευτική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι αηφόρο και βιώσιμο, γιατί αν αδειάσουν οι θάλασσες δεν θα έχουμε τίποτα να ψαρεύουμε. Και δεν ευσταθεί ούτε από οικονομική ε, πλευράς, ούτε από οικολογική, ούτε αηφόρο είναι, ούτε βιώσιμο. Αυτό το θέμα λοιπόν της επανεθνικοποίησης είναι κάτι που η δική μου πολιτική ομάδα απορρίπτει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τις τροπολογίες για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Ε, κύριε Λαζάρου, θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρα από αυτά που σας είχα πει στις 9 Φεβρουαρίου, δεν έχω τίποτε να προσθέσω. Αλλά είμαι διαθέσιμος για να λύσω τυχόν απορίες. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνεδρίο έχει ως καθήκον να φέρει στην προσοχή των νομοθετικών αρχών οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να σημειωθούν κατά τη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Είμαστε ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι γιατί σας υποβάλαμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε από τους ελέγχους μας με αδιάσυστα στοιχεία, συστάσεις και συμπεράσματα. Δεν είναι δική μας δικαιοδοσία να κάνουμε πολιτικές προτάσεις και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε τη δυνατότητα απλώς να σας τα γνωστοποιήσουμε. Εσείς θα δείτε πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαζάρο. Πραγματικά η έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, επέστησε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα και το θέμα των κολυδηλίων και τώρα ερχόμαστε πολιτικά να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι σωστές πολιτικές ε, επιπτώσεις και τα συμπεράσματα που θα πρέπει να εξαχθούν. Τώρα δεν ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος παρευρίσκεται και ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ συστηθείτε σύντομα γιατί η γραμματεία δεν μπόρεσε να μου δώσει το όνομά σας. Παρακαλώ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Δομένικος Λευγέ. <laughs> Και πρόσφατα διορίστηκα για να παρακολουθώ την εφαρμογή του κανονισμού ΦΕΑΜΠ. Ιδιαίτερα δε τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής Αλληλείας και της Επιτροπής σας. Αυτό που με ρωτάτε τώρα, καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να αντιδράσουμε και θα αρχίσω πολύ σύντομα να σχόλιά μου στο 12 και το 13 που αφορά την επανεθνικοποίηση της ΚΑΛΠ που ζήτησε ένα, μια βουλευτής. Για τις τέσσερις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα τις αναφέρω ανάποδα. Δηλαδή, από το πιο βραχυπρόθεσμο μέτρο μέχρι το πιο μακροπρόθεσμο. Η πρώτη σύσταση αφορά την ενημέρωση του Μητρώου των Λιαρίων, του νιολογίου που λέμε. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η τακτική ενημέρωση από τα κράτη-μέλη του νεολογίου είναι κάτι που γίνεται. Και αν ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από το ΦΕΠ δεν έχει ταυτιστεί όπως πρέπει στο νεολόγιο αυτό, τότε θα θεωρείται ανομαλία και ατασταλία και θα διακόπτεται ίσως και η επιχορήγησή του. Δεύτερη σύσταση, λίγο πιο μακροπρόθεσμη, αφορά την εφαρμογή του εξυγχρονισμού του στόλου μας χωρίς να πλήττει όμως την ability του catch fish όπως λέμε εμείς. Εννοούμε βέβαια την... τα ψάρια που βγάζουμε από το νερό, όχι αυτά που βάλουμε στη στεριά, που βγάζουμε από το νερό. Αυτό δεν έχει, δεν έχει ελεγχθεί πλήρως από τα κράτη-μέλη όταν υπέβαλαν τα σχέδια εξυγχρονισμού και το ελεκτικό συνέδριο ταύτισε αυτή την ανομαλία και γι' αυτό η Κομισιόν ανέλαβε ένα σχέδιο δράσης πρότεινε δηλαδή μια νομικός αποδεκτή ερμηνεία του τι σημαίνει αποτελεσματικότητα και όχι μόνο δυνατότητες ή δυναμικό του κάποιου πλοιαρίου και μετά προβλέφθηκε ολόκληρη διαδικασία ελέγχου ώστε να είναι βέβαιον επαλήθευσης ώστε δεν αυξάνεται κατά τον εξυγχρονισμό η δυνατότητα της αλίευσης ενός πλοίου. Και θελήσαμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλα τα σχέδια που εγκρίνονται σέβονται τον όρο αυτό. Αυτή η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Για ορισμένα κράτη-μέλη αυτό απαιτεί τεράστια δουλειά γιατί υπάρχουν χιλιάδες προγράμματα που πρέπει να επαληθευθούν. Άρα και κάποιο κόστος. Τρίτον, η μεταφορά των αλληλευτικών δικαιωμάτων ως προς τον εξυγχρονισμό. Εδώ είναι ακόμα πιο μακροπρόθεσμος ο στόχος. Η εφαρμογή ενός καινούριου ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλληλείας, ακόμη συζητιέται από το Κοινοβούλιο και στοχεύει στο να έχουν πράγματι πρόσβαση οι αλληλείς σε ό,τι πληροφορίες χρειάζονται για τον εξυγχρονισμό και το σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας γιατί όπως γνωρίζετε είναι από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα η θνησιμότητα και τα ατυχήματα είναι πολύ ψηλά και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας για να είναι πιο βιώσιμη η αλλιευτική δραστηριότητα. Τέλος, η μείωση των αλλιευμάτων ή της αλλιευτικής δυνατότητας. Δεν ήταν και μεγάλη επιτυχία αυτό. Η πρόταση του ΦΕΑΜΠ στόχευε στην κατάργηση της δυνατότητας χρήσης κοινοτικών πόρων ή ταμείων για τη μείωση των αλληλευτικών δυνατοτήτων, όπως συστήνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, πού θα καταλήξει το Κοινοβούλιο, η ΠΕΜΠ, θα εξαρτηθεί και από τη σύσταση που θα κάνει η Επιτροπή σας. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για ένα τελευταίο θέμα, το σημείο 13 της έκθεσης της κυρίας Ανδρεάσεν, που προτείνει επανεθνικοποίηση της ΚΑΛΠ και άρα πλήρη απόρριψή της. Θέλω να επιμείνω επί τριών θεμάτων. Πρώτον, η έκθεση του λεκτικού συνεδρίου μιλάει για μία μόνο διάσταση ενός τμήματος της ΚΑΛΠ, δηλαδή τον άξονα 1 στον κανονισμό του ΦΕΠ. Ό,τι αφορά δηλαδή τις επιχορηγήσεις στο στολίσκο και για τη μείωση των υπεραλλιεύσεων και για τις επιχορηγήσεις για τον εξυγχρονισμό και όλες τις άλλες κοινωνικο-οικονομικές βοήθειες του αλληλείς. 4,3 δισεκατομμύρια αντιπροσωπεύει το ΦΕΠ και 1,2 από αυτά δίνεται για αυτόν τον άξονα. Κάτι λιγότερο από 30% δηλαδή. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου λοιπόν αφορά μόνο ένα τμήμα αυτού του 30% και τονίζει ελλείψεις που λήφθηκαν υπόψη στην πρόταση της Κομισιόν για την μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν λέει ότι πρέπει να καταργηθεί ο άξον ένα ή όλο το ΦΕΠ και στην προηγούμενη σας συζήτηση φάνηκε ότι τα προβλήματα ορισμένων διαφορετικών ταμείων δεν καταλήγουν αυτόματα σε κατάργηση ας πούμε της περιφερειακής πολιτικής ή του κοινωνικού ταμείου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι συγκεκριμένα προβλήματα σε έναν και μόνο άξονα της λειτουργίας ενός κοινωνικού ταμείου θέλετε να καταλήξουν σε κατάργηση ολόκληρου του ταμείου και όλων των άλλων διαστάσεων όπου δεν ταυτίστηκαν προβλήματα είτε πρόκειται για τη συντήρηση είτε για τον εξυγχρονισμό, την εμπορία ή τις επιχορηγήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη των περιφερειών όπου ζουν οι αλληλείς, βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη δηλαδή και έτσι όπως θα λέγαμε στα αγγλοσαξονικά θα καίγαμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Δηλαδή υπάρχουν, αν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις, για ένα μόνο τμήμα δεν δικαιολογείται ολική απόρριψη. Θα ήθελα εδώ να επιμείνω ότι στο ότι δεν πρέπει να αγνοούμε ότι μια επανεθνικοποίηση της ΚΑΛΠ θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση όπως υπήρχε προηγουμένως ως προς τις επιχορηγήσεις για την αύξηση του δυναμικού ή της αλληλευτικής ικανότητος. Oui, beaucoup. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που έχει σημασία και αποφασιστική είναι να βεβαιωθούμε εδώ στην Επιτροπή μας για το εξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να πιάνουν τόπο να είναι όσο γίνεται πιο χρηστή και φιδωλή η διαχείρισή τους και στοχευμένη. Αυτή είναι η βασική μα ανησυχία και το μέλημα. Τώρα για τους στόχου της πολιτικής, ποιοι είναι οι σωστοί στόχοι, ε, μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη διάφορες πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι σαφέστατο. Και αυτό που ανέφερε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευσταθεί και συνηγορεί υπέρ της ε, κοινοτικοποίησης ορισμένων πολιτικών. Μα αυτό ήτανε και βάση για τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως και συνάδελφοι που διαφωνούν με αυτή την αντίληψη. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι οι προτάσεις του Αλλακτικού Συνεδρίου για πιο φιδωλή και χρηστή διαχείριση ε, θα πρέπει να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ενεργά και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη γιατί όπου επισημαίνονται ελλείψεις, δυσκολίες και δυσλειτουργίες θα πρέπει το συντομότερο να διορθώνονται και αυτό είναι προς το κοινό όφελος όλων των ενεχομένων. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια τώρα για να οπλώσει η κυρία Ανδρέζεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σχόλια που έκανε ο κ. Γκάιερ. Είπε ότι είναι αντίθετος με την επανεθνικοποίηση διότι έτσι στόλοι θα μπορούσαν να επεκταθούν, να αυξηθούν και θα λιεύαμε όλα τα ψάρια του ωκεανού. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν έχουμε αφήσει λέπη. <laughs> Ξέρετε ότι η επανεθνικοποίηση δεν θα χειροτερεύσει την κατάσταση. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε κοινή αλληλευτική πολιτική και τα κράτη-μέλη εφάρμοζαν τη δική τους αλληλευτική πολιτική. Και λειτουργούσε καλά. Γιατί πρέπει να ανταλλάξουμε αυτό το σύστημα και να βάλουμε κάποιο άλλο που δεν λειτουργεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται σε μία πτυχή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που είναι αληθές με ένα προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού για την αλληλευτική πολιτική και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν λέγει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία καυγαλαία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε. 90% των αλευτικών αποθεμάτων υπεραλλιεύονται, 30% από αυτά ε, είναι πάνω από τα βιολογικά όρια τα κανονικά, πάνω από 100.000 θέσεις ε, εργασίας έχουν απολεστεί Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία για να απαλλαγούμε από αυτή την πολιτική. Και όλα αυτά στα πλαίσια της απαλλαγής. Και η απαλλαγή εξετάζει το, στέφεται προς το παρελθόν, όχι το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πολλές απαντήσεις που θεωρούν ότι η νέα λευτική πολιτική θα μας δώσει μια λύση. Τώρα κρίνουμε το παρελθόν και βάσει του παρελθόντος πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση. Υποσχέσεις παραμένουν πάντα υποσχέσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ανδρέασεν. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και ολόκληρη η ημερήσια διάταξη του σημερινού πρωινού. Σας παραπέμπω στην ακρόαση του απογεύματος για τη μελλοντική εργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόπτε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε με την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ.